τρίτη, την τρίτη συνεδρίαση υπό τη νέα θητεία της Επιτροπής Απασχόλησης. Μπορείτε να μιλήσετε και να ακούσετε όλες τις γλώσσες, με εξαίρεση τα φιλανδικά και τα κροατικά, τα οποία δεν είναι γλώσσα της Επιτροπής Απασχόλησης. Σημείο 2. Μερικοί από εσά αναρωτιούνται τι συνέβη με τον πρόεδρο Δυστυχώς ο κύριος Χέντελ, ο πρόεδρος της Επιτροπής, ασθενεί και δεν θα μπορέσουμε δεν θα μπορέσει να πάρει μέρος στις συνεδριάσεις για ένα-δύο μήνες. Θα τον αντικαταστήσω και ελπίζω σύντομα να αναρρώσει και να έρθει και πάλι. Για τον λόγο αυτό λοιπόν βρίσκομαι σε αυτή τη θέση Θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, μόνο ότι δεν είχα τη δυνατότητα να προετοιμαστώ επαρκώς. Σε κάθε περίπτωση θα συνεργαστούμε και ελπίζω να τα καταφέρουμε. Ανακοινώσαμε ότι θα βγάλουμε μια οικογενειακή φωτογραφία όλων των μελών της Επιτροπής όταν επιστρέψει ο κύριος Χάντελ, τότε θα βγάλουμε και την φωτογραφία. Δεν υπάρχει καμία απολύτως διασύνη. Και με αυτόν τον τρόπο περάσαμε στο τρίτο σημείο της ημερησίας διάταξης που αφορά τον πιο αποδοτικό τρόπο εργασίας μας με τη βοήθεια των ηλεκτρονικών ε, διαδικασιών. Στην ουσία καταργήθηκαν τα έγγραφα, γίνονται όλα, ηλεκτρονικά. Θα ήθελα τώρα να σας παρουσιάσω την ομάδα που θα μας πει τι ακριβώς θα πρέπει να κάνουμε σε αυτόν τον κόσμο χωρίς έγγραφα. Δεν θα υπάρχουν λοιπόν τυπωμένα έγγραφα των συνεδριάσεων. Θα πρέπει συνεπώς να επικεντρωθούμε περισσότερο στους υπολογιστές μας. ήθελα να καλέσω την κυρία Χουμπικέ και τη Μηματάρχη και τον κύριο Ντάνινα Γουάντι που είναι υπεύθυνο προγράμματο από τις υπηρεσίες του ίντερνετ να μας πούν πώ ακριβώς θα λειτουργήσει αυτό το σύστημα. Και βεβαίω μπορούμε μετά να θέσουμε και ερωτήσεις. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Το όνομά μου είναι Κιούκεν, ο συνάδελφός μου βρίσκεται στο άλλο μέρος της αίθουσας. Δυστυχώς με τα καλώδια υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα και χρειάστηκε να του ζητήσω να καθίσει στην άλλη πλευρά της αίθουσας. Θα μπορέσουμε να σας δείξουμε στην οθόνη ορισμένα πράγματα. Υπήρχε ένα πρόβλημα με το καλώδιο εκεί, γι' αυτό εγώ βρίσκομαι εδώ. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μας δώσατε να σας μιλήσουμε για τις ή συνεδριάσεις, ηλεκτρονικές συνεδριάσεις. Είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζουμε κάτι τέτοιο στην Επιτροπή και αποτελεί και ένα πείραμα. Όπως είπε και η πρόεδρος καταργούνται τα έγγραφα. Δεν λάβατε κανένα έγγραφο για τη συνάντηση αυτή και δεν θα λάβετε και αργότερα. Είναι μια καινούρια κατάσταση, ένας νέος τρόπος εργασίας. Αυτό που κάνει τώρα το Κοινοβούλιο είναι ότι παρέχει μια ηλεκτρονική εφαρμογή. Η εφαρμογή αυτή ονομάζεται e meeting και εκεί μπορείτε να ανατρέξετε για να βρείτε όλα τα έγγραφα των συνεδριάσεων. Τα έγγραφα είναι πολύ σημαντικά για όλους, ιδιαίτερα για τις επιτροπές και θα πρέπει να τα έχουμε στη διάθεσή μας το συντομότερο δυνατόν και με κάθε τρόπο. Αναπτύξαμε αυτή την εφαρμογή εδώ στο Κοινοβούλιο έτσι ώστε να ανταποκρίνετε στις ανάγκες σας όσο γίνεται περισσότερο. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο e-meeting με το Wi-Fi ή με την κάρτα SIM οπουδήποτε, οποιαδήποτε χρονική στιγμή, σε οποιοδήποτε λάπτοπ, τάμπλετ, smartphone, υπολογιστή, notebook και βεβαίως στην επιφάνεια εργασίας. Διανύμαμε μόνον ένα έγγραφο, το βρείτε μπροστά σας, στα έδρανά σας. Εν περίληψη βλέπετε πώς μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στο e-meeting. Βλέπετε λοιπόν τι μπορείτε να κάνετε για να έχετε πρόσβαση με το δικό σας, τη δική σας συσκευή. Με την άδεια της Προέδρου θα ήθελα να, αναπαρακαλέσω παρακαλέσω το συνάδελφό μου να σας πει λεπτομερέστερα πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα αυτή η εφαρμογή του e-meeting. Εφαγητό. Η εφαρμογή e-meeting είναι μία ε, εφαρμογή που βασίζεται στην ιστοσελίδα, στο web, δεν χρειάζεται δηλαδή να εγκαταστήσουμε τίποτα για να το χρησιμοποιήσουμε. Σημαίνει επίσης ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε συσκευή, desktop, επανεργασία, iPad κτλ. Για να έχετε πρόσβαση στην εφαρμογή, πληκτρολογείτε και σας παρακαλώ να το κάνετε αν θέλετε, www.europal, και μετά κάθετος e-meeting. Επειδή είναι εσωτερική η εφαρμογή, δηλαδή μόνο οι εργαζόμενοι για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα άτομα δηλαδή που είναι εγγεγραμμένα στο σύστημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν δικαίωμα πρόσβασης. Γράφω λοιπόν το όνομα χρήστη εδώ και βάζω και τον κωδικό πρόσβασης, τον κλειδάριθμο. Α, με αυτόν τον τρόπο θα δείτε όλοι τον κλειδάριθμό μου. Περνάμε από τη δική μας πύλη, αυτή είναι η ιστοσελίδα του EPNET, από την οποία έχουμε, στην οποία έχουμε όλη πρόσβαση. Την πρώτη φορά που μπαίνετε έχετε μία οθόνη που σας εξηγεί ότι θα πρέπει να ακολουθήσετε ορισμένα βήματα. Θα πρέπει να επιλέξετε την ε, γλώσσα την επιτροπή, και την επιτροπή. Στην αριστερή πλευρά βλέπετε τη γλώσσα. Μετά έχετε την επιτροπή. Το e-meeting μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε επιτροπή. Για παράδειγμα, ας πούμε στην Επιτροπή Employment, απασχόλησης. Το σύστημα δίνει όλες τις πληροφορίες και παρέχει επικαιροποιημένη πληροφόρηση. Δηλαδή αν κάποιος προσθέσει 3-5 λεπτά κάτι, αυτό θα μπορέσει να ε, απεικονιστεί εδώ. Για δέστε εδώ, στη δεξιά πλευρά βλέπω την ημερησία διάταξη. Βλέπετε τα θέματα της ημερησία διάταξης, βλέπετε και επιπλέον πληροφορίες που αφορούν τον εισηγητή και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτές είναι όλες οι πληροφορίες που συνήθως παρέχονται σε έντυπη μορφή σε όλες τις επιτροπές. Στην δεξιά πλευρά έχω τα έγγραφα, είναι περίπου το ίδιο, αλλά εστιάζεται η προσοχή στα έγγραφα. Δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο είναι εύκολο να έχει κανείς πρόσβαση στα έγγραφα άμεσα από αυτή τη σελίδα. Μπορώ να δω σε ποια γλώσσα διατίθενται τα έγγραφα. Αυτό ισχύει για όλα τα έγγραφα. Ας δοκιμάσω να ανοίξω ένα έγγραφο, ας πούμε αυτό το σχέδιο νομοδότης, κλικάρω και ανοίγει το έγγραφο. Μπορώ λοιπόν να έχω άμεση πρόσβαση στο έγγραφο εδώ και σε περίπτωση που θα ήθελα να υπάρχει μια λιλεπίδραση, μπορώ να το ανοίξω σε μια ε, τρίτη εφαρμογή. Μπορώ να το ανοίξω ε, εδώ και να κάνω, να σχεδιάσω, να πω ότι αυτό το θέλω, να το υπογραμμίσω, δηλαδή να παρέμβω άμεσα στο έγγραφο. Αυτό είναι το δικό μου έγγραφο, εδώ μπορώ να αναφέρω ότι έχω κάνει αλλαγές, δηλαδή να το χρησιμοποιήσω ως σημειωματάριο. Κάνω τις αλλαγές και μετά πατάω το save. Ας πούμε εδώ μπορώ να το τονίσω, εδώ μπορώ να το διαγράψω. αυτό είναι ένα αντίγραφο του εγγράφου, αλλά είναι δικό μου. Κανένας ε, δεν θα έχει πρόσβαση σε αυτό θα αφορά μόνο τη δική μου επιφάνεια εργασίας. Και μόλις γίνουν όλες αυτές οι αλλαγές, αυτό θα πρέπει να κάνετε. Κάνετε αυτό που κάνετε με ένα στυλό. Μπορείτε εύκολα να το μοιραστείτε με κάποιον άλλον. Μπορώ να το στείλω με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, να το στείλω στα μέλη και να στείλω κάποια κοινοποίηση στον βοηθό αυτός που ελάβει αυτό το έγγραφο θα το λάβει με όλες τις σημειώσεις και τις πληροφορίες που έχουν προσθεθεί στο συγκεκριμένο έγγραφο. Αυτό είναι μια κλασική περίπτωση του e-meeting. Αυτό μπορεί να γίνει για οποιαδήποτε εφαρμογή. Μπορώ να περάσω σε μια άλλη επιτροπή. Είναι ενδεχόμενο τα μέλη, ένα μέλος να παρακολουθεί δύο επιτροπές σχεδόν παράλληλα. Μπορεί λοιπόν να συνεχίσει να εργάζεται με βάση τα έγγραφα μιας άλλης επιτροπής. Για παράδειγμα μπορώ να κλικάρω στο τζούρι και εκεί να πάρω όλες τις πληροφορίες που αφορούν τη συγκεκριμένη επιτροπή. Αυτή είναι η εφαρμογή που υποτίθεται ότι θα αντικαταστήσει το ντοσιέ UNICA, δηλαδή τα έγγραφα που τυπώνονται κάθε φορά. 20 εκατομμύρια σελίδες το χρόνο τα 20 εκατομμύρια σελίδε σελίδες θα αντικατασταθούν με το, e, ε, από το e-meeting. Όταν είμαι σε μια επιτροπή, εδώ όπως βλέπετε, έχω μια άλλη ενδιαφέρουσα εφαρμογή που λέγεται e-committee. Αν κλικάρω στο e-committee θα περάσω απευθείας στο intranet της ιστοσελίδας της επιτροπής. Με το intranet εννοώ ότι ε, έχουμε μια ιστοσελίδα με πλήρη πληροφόρηση σχετικά με το έργο των επιτροπών. Εγώ βεβαίως έχω πρόσβαση από το εξωτερικό Wi-Fi, αλλά ε, χρειάζεται κάποιος χρόνος. Σε κάθε περίπτωση, σε όλα αυτά μπορείτε να έχετε πρόσβαση από την επιφάνεια εργασία σας. Απαιτείται κάποιος χρόνος. Εδώ αποφάσισα να μπω στο ζούρι, μπορώ να το κάνω και για το, την ιστοσελίδα του ε, ίντρανετ. Μισό λεπτό χρειάζεται λίγος χρόνος. Αυτή είναι η ιστοσελίδα του ίντερνετ που έχει όλες τις πληροφορίες. Υπάρχουν 22 ε, ε, ιστοσελίδες εδώ, για παράδειγμα, μπορώ να έχω πρόσβαση σε σχέδιο εκθέσεων στα μέλη. Δηλαδή το website του e-committee είναι πολύ πιο πλήρες. Και εδώ μπορεί κανείς να βρει επιπλέον πληροφορίες. Παρόλα αυτά, για, την, για το e-meeting θα έχετε πληροφορίες που αφορούν μόνο τη συγκεκριμένη ημέρα. Εδώ, για παράδειγμα, μπορώ να έχω πρόσβαση σε όλες τις εκθέσεις. Για κάθε έκθεση υπάρχουν ταμπέλες, υπάρχουν έγγραφα στις διάφορες γλώσσες. Όταν υπάρχουν, γιατί ε, μπορώ να έχω πρόσβαση στο λέγε και να δω ποιος είναι ο κύκλος ζωής του εγγράφου. Κατά βάση έχετε δύο βασικέ προεφαρμογέ, το e-meeting και το e-committee. Αυτά λοιπόν είχα να σας πω σχετικά με τα θέματα αυτά. Εάν έχετε κάποια ερώτηση, είμαι στη διάθεσή σας. Λοιπόν, αν έχετε ερωτήσεις, παρακαλώ. Αλλιώς, μπορούμε να απαντήσουμε σε ερωτήσεις σας και μέσω email και τηλεφωνικά βέβαια. Είμαστε στη διάθεσή σας και με τις δύο αυτές οδούς. Και αν θέλετε, μπορούμε να οργανώσουμε και συνεδριάσεις ενημέρωσης ή και δημερίς. για κατάρτιση για να συνηθίσετε να χρησιμοποιείτε αυτές τις εφαρμογές που θα τις χρειαστείτε κατά την επόμενη λοιπόν αυτή θητεία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Κιόκιο και κύρια Βάντι. υπάρχουν ερωτήσεις. Παρακαλώ. Μία ερώτηση για τον κωδικό. Βεβαίως μπορούμε να φτιάξουμε τα δικά μας, ε, τους δικούς μας κωδικούς, αλλά υπάρχουν ε, ελάχιστες προδιαγραφές, πόσα γράμματα, πόσα νούμερα, κεφαλαία, μικρά. Θα ήταν χρήσιμο να ε, επιλύσουμε και αυτό το θέμα. Ποιες είναι οι ελάχιστες απαιτήσεις, τι πρέπει να περιέχει δηλαδή ο κωδικός μας. Τι γράμματα, τι νούμερα. Άλλες ερωτήσεις, λέει η πρόεδρος. Όχι. Η κυρία Κόκε. Ευχαριστώ πολύ, λέει η κυρία Κιόκε. Το κανονικό σας κωδικό που χρησιμοποιείτε για όλες τις εφαρμογές εντό του Κοινοβουλίου. Το login που σας έδωσε το Κοινοβούλιο. Ο κωδικός για το login που σας έδωσε το Κοινοβούλιο γενικά ισχύει και για την εφαρμογή e-meeting. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Οπότε, το σημείο 3 της μέρης διάταξη. Έγκριση των πρακτικών. Τις συνεδρίες της 7ης, ε, των συνεδριάσεων 7η και 22ης Ιουλίου. Τα έχετε τα πρακτικά και αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις μπορούν να εγκριθούν. Εντάξει, δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Ωραία, πότε να ψηφίσουμε τώρα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για να ψηφίσουμε το Γενικό Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, όλα τα τμήματα. Λοιπόν, για να δω τα εγγραφά μου τώρα. Υπάρχει πρόβλημα με την ισπανική διερμηνία. Υπάρχει πρόβλημα με την ισπανική διερμηνία. Υπάρχει, είναι εντάξει. Α, λειτουργεί. Λειτουργεί στο κανάλι 8. Στο κανάλι 8 θέλετε να ακούσετε ισπανικά. Όχι. Ναι. it's with... Λοιπόν, αρχίζουμε την ψηφοφορία για το σχέδιο γνωμοδότησης της Μαρίας Αρένα για τον προϋπολογισμό. Παράγραφος 1. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Mm -hmm. Παράγραφος 1α. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 1b. Τροπολογία 4. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος. Στην παράγραφο 1α τροπολογία 3. Υπέρ παρακαλώ κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 1b. Για την τροπολογία 5 έχει ζητηθεί κατά τμήματα ψηφοφορία. Το πρώτο τμήμα. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά Λοιπόν, ας ελέγξουμε παρακαλώ. Έχετε τις ηλεκτρονικές σας κάρτες. Παρακαλώ ψηφίστε. Ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα. Υπέρ κατά ή αποχή. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε ψηφοφορίες. Λοιπόν, εγκρίνεται. Το τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Το τέταρτο τμήμα υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. Καλά. Καλά. Να ελέγξουμε. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά το τέταρτο τμήμα. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Στην παράγραφο 1c υπέρ κατά Αποχές. Δεν είναι σαφές. Να ελέγξουμε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Α, αμφίροποι. Αλλά εγκρίνεται. Παράγραφος 2. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτε. Τροπολογία 8 στην παράγραφο 2α Κατά τμήματα ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Στην παράγραφο 3, τροπολογία 9. Υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. Στην παράγραφο 3 πάντα τροπολογία 10. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Στην παράγραφο 3 πάντα, τροπολογία 11. Με μία προφορική τροπολόγηση. Αν δεν έχετε αντιρρήσεις στην προφορική τροπολόγηση. Υπάρχουν άλλοι που να έχουν αντίρρηση παρακαλώ. Α, υπάρχουν. Είναι πάνω από τρεις. Οπότε η προφορική τροπολόγηση ε, δεν μπορεί να γίνει δεκτή. Θα ψηφίσουμε το αρχικό κείμενο. Χωρίς προφορική τροποποίηση. Υπέρ παρακαλώ, υπέρ. Κατά παρακαλώ. Άποχες. Απορρίπτεται. Τροπολογία 12 στην παράγραφο 3. Υπέρ. Μ, κατά. Αποχές. Δεν ήταν σαφές ε, να ελέγξουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Στην παράγραφο 3α. Τροπολογία 13. Υπέρ. Κάτω. Αποχές. Εγκρίνεται. Καλά. Ίσως να μην ήταν απόλυτα σαφές, οπότε να ελέγξουμε. Και εδώ, ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Στην παράγραφο 3α, τροπολογία 14. με προφορική τροποποίηση. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Στην παράγραφο 3β, τροπολογία 15, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 3Β Τροπολογία 16 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 4. Τροπολογία 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Μία προφορική τροπολόγηση. Α, με συγχωρείτε. Α, όχι, όχι, αποσύρεται. Καταπίπτει. Καταπίπτει. Τροπολογία 18. Ποιοι είναι υπέρ Τις πρώτου τμήματος τη Τροπολογία 18. Κατά αποχές. Πρέπει να ελέγξουμε. 18 πρώτο τμήμα. Αυτό ψηφίζουμε τώρα. Ψηφίσατε όλοι. Ευχαριστώ πολύ. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Α, καλά, ελέγχουμε. Ψηφίσατε όλοι. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, είχατε δίκιο. Απορρίπτεται. Παράγραφος 4, τροπολογία 19. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Πρέπει να ελέγξουμε. Ψηφίσατε όλοι. Εγκρίνεται. Παράγραφος 5, τροπολογία 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 6. Τροπολογία 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 6. Τροπολογία 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 6α, τροπολογία 23, υπέρ, κατά, αποχές πρέπει να ελέγξουμε. Ψηφίσατε όλοι. Υπάρχει ένας αναπληρωματικός παραπάνω που ψηφίζει από την ομάδα των σοσιαλιστών. Εντάξει. Ωραία. Για να το αποτέλεσμα. Απορρίπτεται. Στην 6α τροπολογία 24, 25. Υπέρ. κατά αποχές. Πρέπει να ελέγξουμε και αυτήν. I made Συγχωρείτε, έκανα λάθος. Ψηφίζουμε την τροπολογία 24. 24. Θα αρχίσουμε πάλι από την αρχή. Ποιοι είναι υπέρ της 24. Κατά και αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα ε, περνάμε στην 25. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές πρέπει να την ελέγξουμε. You have all voted now. Okay. all όλοι. Και τώρα να ψηφίσουμε το σύνολο του σχεδίου γνωμοδότησης όπως τροποποιήθηκε, ονομαστική ψηφοφορία. Άρα θα πρέπει να είναι σαφές. Ποιοι είναι υπέρ. Okay. The vote is closed. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 36 υπέρ, 9 κατά και δύο εποχές. Ευχαριστώ πολύ. Uh, and now it's this. Now it's the vote on the budgetary amendments. Yes. Mm -hmm. Now we'll proceed to the budgetary amendments. Τώρα έχουμε τις τροπολογίες το προϋπολογισμό. Τροπολογία 6500. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. ελέγξουμε το αποτέλεσμα. Ψηφίσατε όλοι. All voted. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφορίες. Διαπιστώνετε ε, ε, Διαπιστώνεται ότι η τροπολογία 6501 απορρίπτεται. Τροπολογία 6502 υπέρ. Κατά. Αποχές. Κατά. Ε, εγκρίνεται, συγγνώμη. Τροπολογία 6502 υπέρ. Κατά. εποχές Εγκρίνεται. Ελεκτρονικός έλεγχος για το 6502. Have all voted. Ψήφισαν όλοι. Oh Η 6503 καταπίπτει για την κρίση 6502 και πάμε στο 6504. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονικός έλεγχος. You have all voted. Thank you. Ψήφισαν όλοι, σας ευχαριστώ. Εγκρίνεται. 65-05. Καταπίπτει. Και πάμε στο 65-06. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 65-07. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 65-08. Πρώτα πρώτα, όσον αφορά τα στοιχεία, πήγαινε υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. έχουμε την προφορική τροπολογία. Ενίσταται κανείς όσον αφορά την προφορική τροπολογία. Όχι, Επομένως θα ψηφίσουμε την προφορική τροπολογία. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συνταπέντε μηδέν Υπέρ. Κατά. Αποχές. Με ηλεκτρονικό έλεγχο. Ψηφίσατε όλοι. Ευχαριστώ. Εγκρίνεται. 65-10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 65-11. ψηφισουμε την 65-11. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 65-12. Υπέρ. αποχες Αποχές. Εγκρίνεται. 65-13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έτσι δεν είναι. Όχι. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. 65-13. Ψηφίσατε όλοι, ευχαριστώ. Απορρίπτεται. 65-14, υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα καθόλου και επομένως θα πρέπει και επί του προκειμένου να κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Ψηφίσατε όλοι. Ευχαριστώ. Εγκρίνεται. Στην 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. 65-16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 65, 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 65, 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Πρέπει να γίνει έλεγχος επί του 65-18. Ψηφίσατε όλοι. Εγκρίνεται. Με ένα ψήφο διαφορά και πάμε στο 65-19. Καταπίπτει. 65-20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Κάποια ένσταση σε σχέση με την προφορική τροπολογία. Όχι. Επομένω, ψηφίζουμε την προφορική τροπολογία. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα γίνει έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Απορρίπτεται. 65-21. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Και απορρίπτωτο. Ηλεκτρονικός έλεγχος επί του 65-21. Ψηφίσατε όλοι. Α, είναι τον τίτλο αυτό που νομίζαμε, διότι εγκρίνεται. Και πάμε στο 65-22, το οποίο καταπίπτει, άρα 65-23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Α, απορρίπτεται. 65-24. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. αποχές, εγκρίνεται. 25, υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι, σας ευχαριστώ. ε, κάποιο αναπληρωματικό μέλος θα πρέπει να αποσύρει την ψήφο την οποία έριξε. Έρχεται από τους σοσιαλιστές. Α, εντάξει, τώρα είναι σωστά. Και η τροπολογία απορρίπτεται. Πάμε τώρα στο 65-26. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 65-27. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 65-28. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 65-29. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. 25-29. Ψηφίσατε όλοι. Σας ευχαριστώ. Ε, και εγκρίνεται με διαφορά μιας ψήφου, το οποίο είναι δυσδιάκριτο. vote on 6532. 65-32. Ποιοι είναι υπέρ για το 65-32. Γιατί το 65-30 και 65-31 έχουν καταπέσει, γι' αυτό πήγαμε κατευθείαν στο 65-32. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. 6532 32 Ψηφίσατε όλοι. Ευχαριστώ. Εγκρίνεται. Σε 5.33 καταπίπτει, οπότε πάμε στο 65.34. 65.34. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά. Αποχές απορρίπτεται. 65-35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 65-36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 65-37 Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 38. Δεν επιδέχεται ψηφοφορία. Και πάμε στο 65-39, αλλά ούτε αυτό θα τεθεί σε ψηφοφορία. Πώς είπατε. Α, μάλιστα πάμε κατευθείαν στο 65-41. Εδώ ψηφίζουμε μόνο τα αριθμητικά στοιχεία, τα νούμερα τέλο πάντων. Υπέρ, κατά, αποχές και απορρίπτωτο. 65, 42. Και εδώ ψηφίζουμε μόνο τα στοιχεία. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. απορριπτωται 65, 43, ούτε αυτό θέλει σε ψηφοφορία και πάμε στο 65, 44, ούτε αυτό, πάμε 65, 45. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και τώρα. Έχουμε προφορική τροπολογία από την εισηγήτρια. Έχετε κάποιες ενστάσεις. Όχι. Οπότε ψηφίζουμε. Προφορική τροπολογία. Σε σχέση με υψηλότερα ποσά όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών και υποχρεώσεων. Υπέρ. Κατά. Αποχές. και απορρίπτεται. 65-46 η οποία καταπίπτει και θα ψηφίσουμε την 65-40 θα ψηφίσουμε επί της 65-46 λέει πρόεδρος και ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 65-47 Πρώτα πρώτα για τα ποσά υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Επί των παρατηρήσεων. Πάντα στην 65-47 είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 65-48. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 65-49. Υπέρ. Κατά. Αποχές. ηλεκτρονικός έλεγχος. Χρησιμοποιήστε τι κάρτες ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι και απορρίπτωτε. 65-50. Υπέρ. Κατά. Αποχές. και επ' αυτού ηλεκτρονικό έλεγχο. Ψηφίσατε όλοι και απορρίπτεται. 65-51. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 6552 δεν τη δίδεται ψηφοφορία. Ολοκληρώσαμε όσον αφορά αυτό το σχεδιακημένο για τις τροπολογίες για τον προπολογισμό. Yes, and we will on that. Uh, we proceed. Uh, Συνεχίζουμε την ψηφοφορία για το την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Ψήφι υπέρ. Μισό λεπτό καλύτερα να το κάνουμε ηλεκτρονικά. Ψήφι υπέρ. Ψήφι κατά. Ε, Όχι, εγκρίνεται, εγκρίνεται. Πέρα ψηφοφορία. Θα ψηφίσουμε την κινητοποίηση του εργοκότου ορμήν προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση, τεχνική βοήθεια. Ψήφι ή πέρα. Ναι, ναι, ναι. Ε, έναρξη τη ψηφοφορία. Ψηφίσαμε όλοι, ψηφίσατε όλοι. Εγκρίνεται. Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, Ρουμανία, ψηφίσαμε και γι' αυτό. Ψηφίσατε όλοι. Εγκρίνεται. Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Αραγωνία, Ισπανία. Ψηφίσατε όλοι. Να δούμε μισό λεπτό το αποτέλεσμα. Εγκρίνεται. Ψηφορεί την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για την Ολλανδία. Ψηφίσαμε και γι' αυτό. Πέρασε ψηφοφορία, εγκρίνεται. Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση για την περιοχή της Καστήλια Ιλεών στην Ισπανία. Ψηφίζουμε. Ψηφίζατε όλοι και εγκρίνεται. Πράγμα που σημαίνει ότι τελείωσαν οι ψηφοφορίες. Σας ευχαριστώ που προσθετήκατε για να με βοηθήσετε στην εκπαίδευσή μου. Την επόμενη φορά θα είναι πιο εύκολα τα πράγματα. now reached uh, Περνάμε τώρα στο σημείο 11, Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για το Συντονισμό των Οικονομικών Πολιτικών Υλοποίηση των Προτεραιοτήτων για το 2014. Επιτρέψτε μου να δώσω το λόγο στον κύριο Πριέτο, τον εισηγητή. Κύριε Πριέτο, έχετε το λόγο. Παρακαλώ. Sí, Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο εισηγητής. Κυρία Πρόεδρε. Έχουμε συντάξει αυτή την πρώτη γνωμοδότηση και αυτή τη φορά σας υπενθυμίζω ότι στο πλαίσιο αυτού του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου η Επιτροπή Απασχόληση. τον Φεβρουάριο επί τη αναπτύξεω συνέταξε μια έκθεση ακριβώς όπως και η Οικονομική Επιτροπή. Όμως, όμως όταν φτάσουμε στο σημείο των συστάσεων ανά χώρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την ε, γνωμοδότηση αυτή θα την ε, αναπέμψουμε στην Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 54 του Κανισμού που είναι η κυρίω ομάδια επιτροπή αυτή η οικονομική. Οπότε θα δούμε τώρα τι γίνεται. Είχαμε την συγκρότηση σώμα του Κοινοβουλίου και στα πλαίσια αυτά ε, υπό κάποιες ιδιότητε συνθήκε έπρεπε να συντάξουμε αυτή την οικονομοδότηση. Τέλος πάντων, πέραν αυτού θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να έχουμε έναν αξιόλογο οικοδομικό καλύτερο διάλογο με την υπόλοιπη ομάδα για να είναι οικοδομητική αυτή η γνωμοδότηση και τόσο για να αξιολογηθούν τα τα μνημόνια αναχώρα τα οποία έχει εγκρίνει το Συμβούλιο. Απλώς είναι μια απόπειρα για να προσπαθήσουμε να επηρεάσουμε ε, το, την επόμενη έκθεση που θα γίνει για την ανάπτυξη και τον κόστος αυτής που θα γίνει την επόμενη γιατί ο, ο μιλητής θεωρεί ότι θα πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές κάποιες αλλαγές ήδη έχουν ανακοινωθεί και είπαμε ότι ε, συγκεντρώνει τη Γενική Σένεση των κομμάτων όλων ε, τώρα που θα συγκροτηθεί και η Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχουμε επίσης Αυτά όλα τα οποία συντρέχουν τώρα την νομική συγκύρια, οπότε θα πρέπει να γίνει μεγαλύτερη προσπάθεια και βρισκόμαστε τώρα σε κάποια κρίσιμη στιγμή όσον αφορά αυτή τη διαδικασία, αυτή την πορεία ανάπτυξης και αυτό το μήνα πρέπει να το στείλουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Έχουμε 4-5 χρόνια ε, τέτοιων εξαμήνων και είχαμε πει ότι θα πρέπει σε όλη τη διαδικασία να υπάρξει κάποια δημοκρατική νομοποίηση γιατί δεν έχει νόημα το να αποφαίνεται το Ευρωπαϊκό ε, ε, Κοινοβούλιο για τις Εθνικές Μεταρρυθμίσεις και τον Συστάσεων Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 3-4 μήνες πιο πέρα να έχουμε μια τέτοια έγκριση αυτών χωρίς να λαμβάνει την υπόψη το Κοινοβούλιο γιατί χρειάζεται κάποιο είδους νοημοποίηση αυτής της οικονομικής διακυβέρνησης θα πρέπει με όλα αυτά κάπως να δράζονται περισσότερο στην δημοκρατική νομοποίηση. Ε, γιατί επ' αυτού έχει τη σχετική κυριαρχία, αυτονομία, αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οπότε και εμείς αενάς παραλαμβάνουμε ότι θα πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο και έτσι να παρέχονται κάποιες εγγυήσεις και αυτό να αποτελεί μόνο μια γνωμοδότηση, αλλά είναι κάτι σαν απόφαση ε, του Κοινοβουλίου για όλη αυτή τη διαδικασία. Τι έχουμε σε αυτή την έκθεση. Πρώτα πρώτα αξιολογούμε την κατάσταση και λέμε ότι είναι αλήθεια ότι την τελευταία χρονιά σε σχέση με την προηγούμενη είχαμε κάποιες ελαφρές βελτιώσεις από πλευράς του του, του, του, του εισηγητή σας μακροοικονομικές είναι αυτές όμως βελτιώσεις γιατί στην πραγματική οικονομία εκατομμύρια Ευρωπαίων μαστίζονται όλο ένα και περισσότερο στη συγκεκριμένη οικονομική ζώνη και όλο ένα και τα πράγματα γίνονται σκληρότερα για αυτούς τους, ε, τους Ευρωπαίους ε, οι, οι μισθοί τους ε, έχουμε όλο ένα και περισσότερους μακροπρόθεσμα ανέργους και όλο ένα και περισσότερο πλήσονται οι νέοι σε ανεργία ή σε επισφαλή θέση απασχόλησης. Άρα και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάτι να κάνει. Και αυτό που θα πρέπει να κάνει είναι να πετύχει ότι με ευκαιρία αυτή, αυτή τα καλύτερα μακροοικονομικά με αυτές τις καλές τάσεις να τα επιστατήσει τα καλά στοιχεία, να τα κάνει κάποιες πολιτικές, ούτω ώστε έξω από την κρίση να είναι πιο ξεκάθαρη, πιο γρήγορη. Να έχουμε ανάπτυξη, να μην έχουμε ανισότητες, να μην έχουμε φτώχεια και αυτός είναι ο κοινός Να δοθεί όθηση σε κάποια απασχόληση αξιοπρεπή και διαρκή. Οπότε, επομένως, με αυτό το εξάμεινο, με την ευκαιρία αυτή με την ευκαιρία αυτό της καλής μακροοικονομίας να κάνουμε κάτι μέσα στις αγορές για να βελτιωθεί η ζωή του κοσμάκη. Επομένω, τι θα κάνουμε, πολλά. Ζητήσαμε επανειλημμένα εδώ από την Επιτροπή της Απασχόλησης και η Ολομέλεια του Κοινοβουλίου το ζήτησε. Πρώτα πρώτα, αυτό που είπε και ο κύριος Γιούγκερ. Μία χαλάρωση αυτής της πολύ σκληρής λιτότητας που έχει επιβληθεί με τα προγράμματα προσαρμογής των κράτων μελών. Χτυπιέται έτσι η οικονομία, χτυπιούνται και οι όροι διαβίωση των πολιτών. Άρα, περισσότερη ευελιξία. Να δοθεί μια όθηση στην απασχόληση. Να βοηθηθεί η ανάπτυξη και να έχουμε και ανάπτυξη. Να σταματήσουμε να πνίγουμε την ε, οικονομία. Επίσης, ανακοινώθηκε ότι θα έχουμε κάποιο είδους προγράμματα αξιολόγησης για κάθε μέτρο προσαρμογής και ζητήσαμε οι κοινωνικοί δείκτες να μην αφορούν μόνο τα προγράμματα προσαρμογής, να γίνεται μια αξιολόγηση συνεχής, πάγια, για όλες τις συστάσεις της Κομισιόν προς τα κράτη Και υπενθυμίζουμε ότι η Επιτροπή μας εδώ πάγια το έχει ζητήσει αυτό. Αυτοί οι κοινωνικοί δείκτες να είναι δεσμευτικοί να είναι το ίδιο δεσμευτική όπως και οι μακροοικονομικοί δείκτες. Να μην ξεχνάμε ότι οποιαδήποτε απόφαση για οποιοδήποτε τομέα της οικονομίας θίγει αφορά εκατομμύρια Ευρωπαίων. Άρα θα πρέπει να πετύχουμε και κάτι άλλο. Η απασχόληση να είναι στην καρδιά της πολιτικής αυτής που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό ζητάει το Κοινοβούλιο. Οπότε και για αυτό ζητάμε όταν έρθουν εδώ οι επίτροποι για ακροάσεις να μας πάνε συγκεκριμένα με το χαρτοφυλάκιά τους τι θα κάνουν για να βοηθήσουν την υπόθεση αυτή. 10, 11 έως 11 εκατομμύρια ανέργους έχουμε σήμερα εδώ πέρα. Έχουμε φτάσει σε ρεκόρ για την Ευρώπη. Υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ του τι γίνεται στην Αυστρία και από την άλλη μεριά μεταξύ Ισπανίας και Ελλάδας. Κάτι πρέπει να κάνει η Ευρώπη θα πρέπει να στείλουμε επιτέλους το μήνυμα στον κόσμο ότι κάθε πολιτική ευρωπαϊκή θα έχει βασικό στόχο ακριβώς αυτό, την απασχόληση. Και αυτό να ζητήσουμε από τους επιτρόπους να μας πούν με το χαρτοφυλάκια τους πώς θα βοηθήσουν συγκεκριμένα ούτως ώστε να δοθεί μια τέτοια δυναμική για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Ταυτόχρονα. Τι ζητάμε. Να αποκτήσουμε κάποια μέσα πολιτικής, εργαλεία όπως λέμε, ούτως ώστε να κάνουμε αυτό το οποίο δεν κάνουμε ούτε τη μία χρονιά, ούτε την επόμενη και ούτω καθεξής. Επήγε αυτό. Περισσότερες θέσεις εργασίας για τους νέους. Έχουμε τώρα αυτό το πρόγραμμα της εγγύησης για την νεότητα. Αυτό όμως απλώς έχει μεταφέρει, έχει στείλει κάποιους πόρους στα κράτη-μέλη, αλλά θα πρέπει να πούμε ακριβώς τι χρηματοδοτείται, τι δεν χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Κρούα. Και να δούμε πώς θα πρεκοδοτηθεί ακόμη περισσότερο αυτή η υπόθεση. Και αυτό να γίνει εκμεταλλευόμενη την ευκαιρία των επομένων συναντήσεων κορυφής για να δώσουμε μια λύση σε αυτή την τραγωδία των νέων που πάσχουν από αυτή την ανεργία. Επίση, είναι πάρα πολύ σημαντικό να βελτιώσουμε τη βιομηχανική πολιτική, είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταπολεμήσουμε το κοινωνικό dumping, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Το πώ δημιουργείται αυτού του είδους η φτώχεια σε σχέση με τη δουλειά, την απασχόληση. Ο, ο ΣΑΕ παρουσίασε τις προάλλε μια έκθεση και έλεγε ότι οι περικοπέ μισθού που έχουν γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σε περισσότερη παραγωγικότητα, αλλά επίση έχουν αρχίσει να γίνονται αντιπαραγωγικά αυτά τα μέτρα γιατί τώρα υπάρχει ένα γενικευμένο κλίμα ή αποτέλεσμα ε, που έχει κάνει τον κόσμο πιο φτωχό. Άρα θα πρέπει κάτι να κάνουμε για να είναι πιο αξιοπρεπεί οι συνθήκε διαβίωση των ε, εργαζομένων. Να μην πλησιάζει ο κόσμο ή να μην πέφτει κάτω από το κατόφλι τη φτώχεια, άρα θα πρέπει τα διάφορα αυτά μέτρα να αναθεωρηθούν όποιος επομένως δουλεύει να μπορεί με το μισθό, με την αμοιβή να, έχει το καλάθι τέλο πάντων του καταναλωτή να μπορεί να το γεμίσει, να πληρώνει το τυχόν δάνειο το στεγαστικό που έχει κλπ. κλπ. Γιατί αυτά είναι τα βασικά στοιχεία της ταυτότητας της Ευρώπης. Να βοηθήσουμε νέα προγράμματα, νέα μέτρα για μια προσθεμένη αξία και να σταματήσει αυτού του είδους η μακροπρόθεσμη ενεργεία που είναι η άλλη όψη της τραγωδίας που πλήθ, τους νέους, αλλά εκτός από αυτούς έχουμε και αυτούς τους 45-50 ετών οι οποίοι βγαίνουν από την αγορά εργασίας μετά από αυτά τα 3-4 ε, χρόνια κρίσης που δεν μπορούν να βρουν δουλειά για όλους αυτούς τους λόγους του Ρημοτική Κομισιόν και τα κρατημέλη θα πρέπει να εκμεταλλευτούν αυτή την καινούργια ε, θητεία και σε αυτή την καινούργια φάση Ας δώσουμε επομένως κάποιες πιο ρόδινες προοπτικές στον κόσμο που υποφέρει τόσο πολύ παρά τις μακροοικονομικές βελτιώσεις. Η Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο Σκιώδης συζητητής από την ορμάδα ε, του ΕΛΚ. Βερόνικα Λόπε Φοντάνη. Ευχαριστώ. Και άλλη μια φορά συζητάμε για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εργασία του, για την κατάρτιση αυτές της γνωμοδότησης και είμαι σίγουρη γιατί είναι τρίτη φορά που εργαζόμαστε για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και πιστεύω λοιπόν, είμαι πεπισμένη ότι και αυτή τη φορά θα εργαστούμε θετικά για τα συμφέροντα των πολιτών και την εικόνα του Κοινοβουλίου υπέρ πολλών σημείων που αναφέρει η γνωμοδότηση συγκεκριμένα στις αναφορές που γίνονται στην ανέχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Είναι πολύ επιτυχημένες αυτές οι διατυπώσεις. Α, για άλλα σημεία είμαι λιγότερο σύμφωνη. Όταν ε, θεωρείτε ότι οι πολιτικές που έχουν ακολουθηθεί είναι ε, υπεύθυνε για τη φτώχεια και τη μείωση της κοινωνικής ε, πρόνοιας. Όπως λέει η Κομισιόν, η λιτότητα δεν είναι ο τελικός στόχος. Ήταν μια αναγκαιότητα για να αποφευχθεί η χρεοκοπία κάποιων κρατών μελών και η καταστροφή του ευρώ. Αν δεν είχαν υπάρξει αυτές οι πολιτικές θα ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα. Τώρα λοιπόν οι προβλέψεις είναι ότι για το 2015 θα υπάρξει ανάπτυξη σε όλες τις χώρες, ανάπτυξη του ΑΕΠ. Αυτό είναι πολύ διαφορετικό από το περιβάλλον κρίσης που είχαμε πριν από δύο χρόνια. Συμφωνώ με τον εισηγητή ότι πρέπει να τονίσουμε περισσότερο τις κοινωνικές πλευρές, να επικεντρωθούμε στην ανάπτυξη και την απασχόληση. Αυτό είναι θεμελιώδες για όλους. Αλλά να μην ξεχάσουμε παράλληλα την ανάγκη να υπάρχει έλεγχος ε, των δημοσιονομικών. Πρέπει να μειωθεί το χρέος. Δεν μπορούμε να αφήσουμε να πάνε χαμένες όλες οι προσπάθειες που κάνουμε μέχρι τώρα. Όλες οι θυσίες ε, των πολιτών μας. Τώρα είναι η στιγμή, τα κράτη-μέλη, τώρα που έχουν ε, μεγαλύτερη, μεγαλύτερα δημοσιονομικά περιθώρια, να κάνουμε προσπάθειες για να επενδύσουμε στην ψηφιακή οικονομία, την καινοτομία και ανάπτυξη. Ξέρω ότι θα καταλήξουμε μέσω τροπολογιών, αλλά με ενδιαφέρει ιδιαίτερα το σημείο 21, όπου λέγεται ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να εφαρμόσουν το σύστημα εγγυήσεων για την νεολαία, αλλά να μιλήσουμε για υποχρέωση και να επιβάλλουμε συγκεκριμένες απαιτήσεις θα περιπλέξει πολύ τα πράγματα για τα κράτη-μέλη. Θα είναι δύσκολο να το αποδεχθούν έτσι. Τα 21 επίσης ε, δις που λέγεται ότι πρέπει να, αποχωρη... να... Ε αφιερωθούν στην απασχόληση. Ωραίο είναι να το λέμε, αλλά δύσκολο θα έχουμε ε, τέτοια κονδύλια. Ο πρόεδρος Γιούνκερ λέει ότι θα αυξηθούν πολύ οι Αυτό είναι πιο ρεαλιστικό. Στο 9 λέγεται ότι οι επίτροποι θα πρέπει να θεωρούν προτεραιότητά τους την απασχόληση. Σωστό να το βάλουμε στην έκθεση. Και συγχαίρω τον εισηγητή για αυτό, για αυτή την πρωτοβουλία. Αλλά, αλλά να του ζητήσουμε να έχουν συγκεκριμένες, ε, ε, συγκεκριμένα τμήματα του προπολογισμού, γι' αυτό μου φαίνεται περίπλοκο. Κάτι άλλο είναι το 5 όπου ζητάει δεσμευτικούς ε, κοινωνικούς δείκτες και αναφέρεται επίσης στην ανάγκη για επενδύσεις για την έρευνα και την εκπαίδευση και ότι όλες αυτές οι επενδύσεις θα πρέπει να μην λαμβάνουν την υπόψη για τον υπολογισμό του υπερβολικού ελλείμματος. Πρέπει να το συζητήσουμε στο ιστορικό της ομάδας μου, αλλά δεν νομίζω ότι θα το αποδεχθούμε. Και το τέσσερα, όπου απαιτείται μια, ένας πραγματικός κοινωνικός πυλώνας εντός της είναι πολύ φιλόδοξο. Καλύτερα να πούμε ότι πρέπει να αναπτυχθεί η κοινωνική διάσταση. Αλλά όπως το έχει διατυπώσει ο εισηγητής, δεν ξέρω ε, μήπως θα μπορούσε να το απαλύνει κάπως το 19. Η συναδελφός μου θα μιλήσει για το θέμα αυτό. Εγώ θα ήθελα ο εισηγητής να μας εξηγήσει τι ακριβώς είναι αυτό που λέει να υπάρχει καλύτερο νομικό πλαίσιο για τους διαμεθοριακούς εργαζόμενους. Είναι η έκθεση για τις αποσπάσεις ή κάτι άλλο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία. Ευχαριστώ. Μερικές φορές ε, θα προτιμήσω να χρησιμοποιήσω την μητρική μου γλώσσα, τα σουηδικά. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, η συγκίτρια της ομάδας Αγαπητοί συνάδελφοι, ως νέο μέλος του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής αυτής, χαίρομαι ιδιαίτερα που παίρνω το λόγο για ένα τόσο ενδιαφέρον θέμα που αφορά τις προτεραιότητε του 2014. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον Σέρκιο και θέλω να πω ότι συμφωνώ με τον εισηγητή ότι η οικονομική ανάκαμψη είναι ακόμα ένα πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα. Πολύ σωστά ο εισηγητής υπογράμμισε το γεγονός ότι η ανεργία των νέων παραμένει σε ένα από τα σοβαρότερα μελήματα στην Ευρώπη σε ορισμένες χώρες. Ε, είναι ιδιαίτερα υψηλό αυτό το επίπεδο. Ο εισηγητής αναφέρεται στην ανάγκη για διαρθρωτικές αλλαγές. Θα λέγω ότι συμφωνώ για το γεγονός ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές είναι πραγματικά αναγκαίες. Το βαθμολόγιο αυτό που έχει εισαχθεί είναι πάρα πολύ χρήσιμο και η ομάδα μου δίχως άλλο θα στηρίξει αυτό το αίτημα. Ενδεχομένως θα πρέπει να σκεφτούμε την επαναδιατύπωση σε ό,τι αφορά τους στόχους για να μην αυξηθεί το βάρος για τις επόμενες γενές. Τέλος, πιστεύω ότι θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στην αντιστήχηση των εργασιών και στις δεξιότητες. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας μελλοντικές αγορές, αγοράς, εργα... ε, αγοράς εργασίας. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε τους απαραίτητους μηχανισμούς και να τους διατηρήσουμε. Κατά την άποψή μου, τα δύο σημεία αυτά είναι σημαντικά για να υπάρξουν περισσότερες ευκαιρίες ε, απασχόλησης στους νέους ανθρώπους. Thank you. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Λαμπαγιόρ, επιτρέψτε μου να δώσω το λόγο στο Ζαμπλαμπέρ, το σκιώδη συγητή. Είναι εδώ ο Ζαν Λαμπέρ, παρακαλώ. Α, η Ζαν Λαμπέρ. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλά θετικά στοιχεία στο σχέδιο γνωμοδότησης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον εισηγητή για τα όσα έχει κάνει. Υπάρχουν πάρα πολλά σημεία που μας βρίσκουν σύμφωνους. Πραγματικά καταβάλλεται μια προσπάθεια να συνυπολογιστεί και η κοινωνική και η οικονομική διάσταση. Όπως αυτό αναφέρεται στην παράγραφο 4. Υπάρχουν και ορισμένα άλλα πράγματα που θα θέλαμε να τονίσουμε περαιτέρω. Επίσης, συμφωνούμε σε ό,τι αφορά την υπόμνηση που έγινε με τη στρατη... για την ευθυγράμμιση με τη στρατηγική του 2020, όχι την αλλακτική, το αλλακτικό χρονοδιάγραμμα που σκεφτόμασταν πριν από δύο χρόνια. Βεβαίως θα πρέπει να υποθούν πολλά για την διάσταση της βιωσιμότητας, για, οικολογική... για τα προγράμματα οικολογικής και ψηφιακής ε... Σε πολλές χώρες μέλη Ε, αναπτύχθηκαν εθνικά προγράμματα. Κατά την άποψή μας, στην παράγραφο 33, δεν, είναι, δεν αναφερόμαστε στη μη εμπλοκή των εθνικών εταίρων. Νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη ευαισθητοποίησης από πλευράς εθνικών κοινοβουλίων. Η κοινωνία των πολιτών πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνει κάτι σε αυτό το τομέα. Πρόκειται για ανθρώπους που πλήττονται άμεσα από το πρόγραμμα αυτό και θα πρέπει να έχουν και κάποια συμμετοχή στο αποτέλεσμα. Καταλαβαίνετε με την σημασία των επενδύσεων, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 12 και τη σημασία και τη σταθερότητα μιας στέγης. Η παροχή της στέγης είναι κάτι που θα πρέπει να αναφερθεί και πάλι στο σημείο αυτό. Στο παρελθόν έχουν γίνει πολλά από ιδιαίτερα έμπειρα άτομα και λαμβάνοντα υπόψη αυτό έχω τη βεβαιότητα ότι θα μπορούσε να προκύψει μια πολύ καλή έκθεση από αυτήν την Επιτροπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ρίνια Ρονακάνα από την ομάδα Γκούε, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά την έκθεση αυτή θα πρέπει να πούμε ότι διαβάζεται ευχάριστα και καταφέρει να θίξει σωστά διάφορα προβλήματα. Υπογραμμίσαμε το, τα δημοκρατικά προβλήματα αυτού του μοντέλου καθώς και τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει για τους πολίτες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους. Συχνά πάρα πολλοί άνεργοι, είναι μακροχρόνιοι άνεργοι, δεν έχουν έναν επαρκή μισθό. Σε κάθε περίπτωση έχουμε και ορισμένες επιθυμίες. Ορισμένες χώρες μέλη θα πρέπει να έχουν περισσότερες δυνατότητες να επενδύσουν στον τομέα της κατάρτισης. Σε κάθε περίπτωση θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την έκθεση αυτή την οποία αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία. Ευχαριστώ. Μακιντάιρ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εμείς δεν διορίσαμε κάποιον σκιώδη εισηγητή για αυτή την έκθεση. Ω συντονίστρια θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την γνωμοδότηση Όλοι μας ε, συμφωνούμε σχετικά με τους στόχους. Το πρόβλημα είναι ότι οι ιδέες μας διαφέρουν σχετικά με τον τρόπο επίτευξης αυτών των στόχων. Βασιζόμενοι στην εμπειρία του προηγούμενου κοινοβουλίου, θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά για να κάνουμε κάτι ιδιαίτερα θετικό σχετικά με αυτό. Υπάρχουν τομείς που δεν θα μας ε, ε, βρουν σύμφωνους, Κάτι που είδαμε ιδιαίτερη χαρά, νομίζω στην παράγραφο 15, εκεί που έγινε μια ιδιαίτερη αναφορά στην ε, μερική απασχόληση, στο part-time, ο εισηγητής συμπεριέλαβε τον όρο εκούσια τελοντική εργασία, μη θελημένη. Η μερική απασχόληση είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να επανέλθουν οι γυναίκες στην αγορά εργασίας. Υπάρχουν πάρα πολλοί που θέλουν την μερική απασχόληση και αν αμαυρώνεται συνέχεια η εικόνα της μερικής απασχόλησης ε, πλήττουμε με έναν τρόπο έμεσο αυτούς τους ανθρώπους. Προέρχομαι από μια χώρα που δεν ανήκει στην Ευρωζώνη και νομίζω ότι είναι σημαντικό τα μέτρα αυτά να μην είναι δεσμευτικά για τις χώρες μέλη που δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ. Απλά θα ήθελα να εκφράσω αυτή την επιφύλαξη. Πάνω απ' όλα πιστεύω ότι αυτό που θα πρέπει να κάνουμε σε όλη την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να καταστήσουμε ευκολότερη την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας από πλευράς των επιχειρήσεων. Το είπα ότι η έκθεση αυτή τη Επιτροπή, οι εκθέσει των κοινοβουλίων δεν δημιουργούν θέσει εργασία. Οι επιχειρήσει δημιουργούν θέσει εργασία και ρόλο μα είναι να το καταστήσουμε αυτό όσο γίνεται πιο εύκολο. Δηλαδή να βοηθήσουμε τι επιχειρήσει να ανθίσουν και να δημιουργήσουν θέσει εργασία. Αυτό είναι ένα τρόπο για να μειωθεί η ανεργία και να μπορέσουν οι νέοι να ενταχθούν στην αγορά εργασία. Πραγματικά θα ήθελα να συμπεριλάβουμε αυτή την προσέγγιση εδώ και με μεγάλη ανυπομονησία περιμένω να ακούσω τον σκιώδη συγητή που θα υποβάλει αυτές τις τροπολογίες και θα συνεργαστεί με τις άλλες ομάδες προς επίτευξη ενός καλού αποτελέσματος. Ευχαριστώ. Κύριο Σάιμον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Επετέλεσε πολύ αξιόλογο έργο παρά τις δύσκολες συνθήκες. Με χαρά Μέχρι σήμερα συνεργαστήκαμε μαζί του πάντως. Εξαιρετική η έκθεσή του. Έχω τώρα τα εξή σημεία για τις παραγράφους 8, 9 και 9. Επί του 8. Εκεί αναφέρεται το πόσο θα ήταν καλύτερα να μπορούμε να μετρήσουμε τα ποσοστά απασχόλησης και όχι ανεργιαστό Στο 9. Μιλούμε για ποιοτικές θέσεις απασχόλησης και ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χαράξει κάποια συγκεκριμένα πολύ προγράμματα για την ε, απασχόληση. Βεβαίως και στο 8 μιλούμε για το τι είναι μετρήσιμο ή τι μετρούμε. Δηλαδή να μετρήσουμε τον αριθμό θέσεων απασχόλησης χωρίς να ξέρουμε πόσες ποιοτικέ θέσει εργασία κάνουμε. Γιατί αυτό όμω δεν και σε κάποιε χώρε όπω το Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουμε δημιουργήσει απασχόληση, αλλά ω επιτοπλίστων είναι οίκιστα ποιοτικέ θέσει εργασία αυτέ. Πρόκειται για εκμετάλλευση. Πρόκειται για ε, δουλειέ part-time, για αυτά τα λεγόμενε μηδενικέ συμβάσει εργασία. Οπότε α μην μετρήσουμε την ποσότητα. Αλλά ακριβώ όπω λέει εδώ πέρα να δούμε πώ θα μετρηθούν οι ποιοτικέ εργασίε. Τώρα, η σκιώδη εισηγητρία στις παρατηρήσεις μα ανέφερε στην παράγραφο 19 το ότι θα πρέπει να υπάρξει κάποιο νομικό πλαίσιο για την κινητικότητα των διασυνεργών εργασιών κλπ. κλπ. Ο δε υποψήφιος πρόεδρος της Επιτροπής είχε πει στο Κοινοβουλίο ξεκάθαρα ότι υπόσχεται αναθεώρηση της οδηγίας για την απόσπαση εργαζομένων ρητά καταδίκασε το κοινωνικό ντάμπινγκ. Είναι παράδειγμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγκεκριμένα ανέφερε το ότι θα πρέπει το, όλα αυτά να ισχύουν και όλες τις χώρες, συλλογικές διαπραγματεύσεις και όλα αυτά θα πρέπει νομίζω σε αυτό μας το κείμενο να τα πούμε ξεκάθαρα. Εμείς ως Επιτροπή Απασχόλησης να είμαστε κατηγορηματικοί. Τέτοια προσέγγιση να υιοθετήσουμε. Αυτά να πούμε στην Επιτροπή. Thank you, Madam Morvai. Πρόεδρος, κυρία Μορβάη. Μπορώ να μιλήσω στα Ουγγρικά. Ναι, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον εισηγητή, τον ευχαριστώ, διότι εδώ έχω στα χέρια μου εξαιρετική έκθεση και μιλούμε για κάποιες αξίες, για σύστημα αξιών Βασικά το ερώτημα το οποίο θέτουμε είναι το εξή. Σε τι σύστημα αξιών θα πρέπει να στηρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να έχουμε ως θεμέλιο την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τη δικαιοσύνη. Γιατί υπάρχει και άλλο σύστημα αξιών σύμφωνα με το οποίο υιοθετούμε την ανταγωνιστικότητα με οποιοδήποτε τίμημα σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία, σε ένα σύστημα αδυσόπιτο που όλα υπαγορεύονται από τα πάνω που παρετείται κανείς και από τη δικαιοσύνη και από την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τελικά περί τίνος πρόκειται. Αυτό το οποίο αναδύεται από την έκθεση είναι ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση πολλοί πιστεύουν κάτι το οποίο είδαμε τις ε, συνέπειες παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύουν λέγω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει για να ανταγωνίζεται τον υπόλοιπο κόσμο, να είναι ανταγωνιστική με τον υπόλοιπο κόσμο. Εκεί όπου οι εργαζόμενοι αμείβονται με λίγα δολάρια την ημέρα και με κάποιες συνθήκες εργασίας εντελώς απαράδεκτες. Και όλα αυτά φυσικά έχουν σκοπό τη μεγιστοποίηση του κέρδους. Με αυτούς λένε θα πρέπει να ανταγωνιστούμε. Βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι Έτσι να ανταγωνιστούμε με, τις, με τον υπόλοιπο κόσμο. Με ποιον, με τον τρίτο κόσμο, τις πιο φτωχές χώρες. Τι θα κάνουμε για αυτές τις χώρες ως Ευρωπαϊκή Ένωση. θα πρέπει να στηριχθούμε στο σύστημα αξιών που απετέλεσε την αφετηρία, το θεμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να, τα διλήμματα τα οποία δημιούργησε η έκθεσή σας. Εσείς ως εισηγητής κάνετε μια σαφή επιλογή. Διαλέξατε τη δικαιοσύνη, την αξιοπρέπεια. Το διαλέξατε ξεκάθαρα. Είπατε όχι, δεν θέλουμε την ανταγωνιστικότητα με οποιοδήποτε τίμημα. Δεν θέλουμε να, να συμπιέσουμε συγνώμη ημερομίστια και μισθούς, να δημιουργήσουμε τους φτωχούς εργαζομένους. Δεν θέλουμε τέτοιες συνθήκες. Να, πώς αντιλαμβάνομαι το τι τώρα ισχύει, το τι κυριαρχεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε τώρα και τις λεγόμενες χώρες δεύτερης κατηγορίας. Εγώ είμαι προέρχομαι από την Ουγγαρία, οπότε θέλω να θέσω και κάτι άλλο το οποίο αναδείται αυτή την έκθεση, το ότι έχουμε τεράστιες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών που ανήκουν στην πρώτη κατηγορία και μεταξύ των χωρών που ανήκουν στη β' κατηγορία. Δηλαδή Ευρώπη δύο ταχυτήτων. Ξέρω ότι εσείς ε, δεν επιστατεύσατε τέτοια ορολογία εισηγητά. Εγώ τα λέω αυτά, δεν τα βάζω στο στόμα σας. Όμως, όμως, να, τέτοιων φαινομένων γινόμεθα μάρτυρες. Εγώ ως Ουγγαρέζα αυτά βλέπω. Α, και αλλού, και στην Πορτογαλία. Κόσμο που μεταναστεύει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορεί να βρει δουλειά. Πάει στις πιο πλούσιες χώρες, πιο ευημερούσες. Και πολλές φορές βέβαια τους εκμεταλλεύονται. Πολλές φορές βρίσκουν δουλειές υπό τραγικές συνθήκες, αλλά έτσι είναι τα πράγματα σήμερα στην Ευρώπη. Πάντως επίσης να σας αναφέρω τι ισχύει για μισθούς και αμοιβέ. Έχουμε μεγάλες διαφορές όσον αφορά το τι πληρώνεται στις πλουσιότερες και την άλλη ευρωπαϊκέ χώρε. Να, Ουγγαρία από τη μια, Αυστρία από την άλλη. Μιλάμε για απόσταση 50 χιλιόμετρων μεταξύ δύο πόλεων. Μια εταιρεία έχει ας πούμε γατρική υποκατάστημα στην Αυστρία και εκεί πληρώνει 5 ή 10 φορές παραπάνω από όσο τους Ούγγρους εργαζομένους της ιδίας εταιρεία στην Ουγγαρία. Χρειάζεται ισότητα και μεταξύ εθνοτήτων και μεταξύ των δύο φίλων, αλλά θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των χωρών εδώ μέσα. Δεν είναι δυνατόν να αποδεχόμεθα τόσο εντυπωσιακές μισθολογικές διαφορές. Και όσον αφορά την αμοιβή και όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας. Επίσης, τι άλλο είπε ο εισηγητής. Είπε να αποφύγουμε ακραίες διαφορές και άρα να έχουμε κάποιον ελάχιστο μισθό 60% δηλαδή του μέσου μισθού σε κάθε χώρα. Και αυτό μου τα της θα πρέπει να ισχύει ως εξή. Να μην επιτρέπεται κανείς να πληρώσει λιγότερο από το 60% του μέσου μισθού σε κάποια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Φερρυπίν στα κρατημέλη μελη της Ανατολικής Ευρώπης. Και έτσι, σε κάποια υποκαταστήματα, σε θηγατρικές τέλο πάντων, να μην κερδίζει ο Ούγγρος εργάτης, ο Ούγγρος εργαζόμενος, κάτω από το 60% του μέσου όρου ε, με τον οποίο αμείβεται ο Αυστριακός στην Αυστρία, ο Γερμανός στη Γερμανία. Να τι πάνε να πει ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Παρακαλώ, μην ξεχνάτε συνάδελφοι ότι και αυτό θα πρέπει να είναι ένας από τους στόχους. Μιλάμε για δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια. Παρακαλώ, λάβετε υπόψη αυτά που σας ανέφερα. Πρόεδρος. Μπάλας. Ευχαριστώ. Συγχαίρω τον εισηγητή για αυτά που έγραψε, αυτά που είπε. Κοιτάξτε, πρέπει να καταλαβαίνουμε πως έχει κατάσταση. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και διάφοροι ηγήμονες ε, ε της οικονομίας θεωρούν ότι η μακροοικονομική πολιτική ε, που ακολουθούμε ως Ευρώπη είναι πρόβλημα για ολόκληρο τον πλανήτη. Αν δεν έχουμε ενεργή δημοσιονομική πολιτική οι διαρθρωτικές ε, μεταρρυθμίσεις που κάνουμε μας οδηγούν στην ύφεση και την στασιμότητα. Από αυτή την άποψη, τα 300 δις που ανήγγειλε ο κύριος Γιούνκερ θα πρέπει να δοθούν σύντομα για να αντισταθμίσουν ε, αυτό το φαινόμενο. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο πρέπει να λάβει υπόψη την κατάσταση αυτή. Η έκθεση είναι θαυμάσια διότι γίνεται μάχη ακριβώς επί των δικτών. Γιατί ανάλογα με την ιεράρχηση που θα κάνουμε στους συζητητές ε, θα καθορίσουμε για την κατεύθυνση της πολιτικής μας. Κάποιοι που είναι σκεπτικοί για τα θέματα αυτά θα πρέπει να αναρωτηθούν για τους ε, δείκτες που θα χρησιμοποιήσουμε για την απασχόληση για παράδειγμα ο ε, αριθμός των ωρών της εβδομαδιαίας εργασίας είναι περίπου ίδιος παντού αλλά το ζήτημα είναι πως κατανέμεται άρα θα πρέπει να δούμε τις συνθήκες ε, κατανομής του χρόνου εργασίας αυτού. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Και το να έχει κανείς ε, απασχόληση δεν σημαίνει ότι έχει και ένα επαρκές εισόδημα. Οι δείκτες, ε, οι οικονομικοί και οι κοινωνικοί πρέπει να ιεραρχηθούν σωστά. Είναι λοιπόν πολύ σωστή η πρόταση αυτή από αυτή την άποψη. Όμως, ποιος έχει την εξουσία. Ξέρουμε γιατί αγωνιζόμεθα, αλλά πρέπει να επαναλάβουμε επανειλημμένα ότι το Κοινοβούλιο θέλει να μπορεί να συναποφασίσει για τα θέματα αυτά. Δεν είναι δυνατόν να είμαστε απλώς ε, ε, ένα σώμα που απλώς έχει καλές προθέσεις. Ευχαριστώ η κυρία Γιασλοβιέτσικα. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή για την θαυμάσια δουλειά. Έχει μια ολοκληρωμένη άποψη για το θέμα της απασχόλησης και τα κοινωνικά ζητήματα. Ιδιαίτερα τώρα που αναλύουμε τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Συμφωνώ με την Σνάλφο Βερόνικα Λόπε Φοντέιν και να προσθέσω και εγώ μερικά σχόλια. Συμφωνώ με το σημείο 9 ιδιαίτερα για το επίπεδο απασχόλησης. Αυτή πρέπει να είναι η προτεραιότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να έχει στο σημείο αυτό πολύ φιλόδοξη στρατηγική. Η αύξηση της απασχόλησης, ωστόσο, πρέπει να είναι κυρίως επίπτωση οικονομικής ανάπτυξης. Δεν μπορεί να γίνει μόνο μέσω στρατηγικών. Όλοι οι επίτροποι θα πρέπει να έχουν υποχρεωτικούς στόχους για ε, σχέδια δράσης για την απασχόληση στον τομέα αρμοδιότητάς τους. Μπορεί να μην είναι απόλυτα εφικτά ε, εφικτή η στόχη, αλλά πρέπει να είναι απόλυτα ευαισθητοποιημένη η Επίτροπη για τα θέματα αυτά. Υπάρχουν όμως κάποιες επικίνδυνες τάσεις για την ποιότητα της εργασίας. Υπάρχουν κάποιες ε, τεχνητές τάσεις ε, στη συζήτηση για την απασχόληση. Ξεκινήσαμε τη συζήτηση αυτή και κατά την προηγούμενη θητεία ε, έχει να κάνει με την απόσπαση των εργαζομένων. Είναι περίπλοκο το θέμα αυτό. Πρέπει να βρούμε τρόπους να μειώσουμε την τεχνητή απασχόληση. Η μερική εργασία θα πρέπει να είναι θελοντική γιατί αλλιώς ε, καταργούνται οι ελευθερίες της εσωτερικής αγοράς. Και για το σημείο 20 συμφωνώ ότι οι περικοπές στην εκπαίδευση και την έρευνα δεν είναι σωστές. Δεν είναι μια καλή τάση να υπάρχουν τέτοιες περικοπές και θα ήταν πολύ αρνητικό να υπάρξουν τέτοιου τύπου περικοπές. Πρέπει λοιπόν να αναλύσουμε όλα τα μέτρα που αφορούν την εκπαίδευση, ούτως ώστε να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε μέσω της εκπαίδευσης ε, αποτελεσματικά τη βελτίωση της κατάστασης. Κάποιες άλλες παρατηρήσεις. Για το σημείο 5, υποχρεωτικοί δείκτες για την απασχόληση. Κοινωνικοί δείκτες. Δεν νομίζω ότι είναι η καλύτερη λύση αυτή. Διότι οι αγορές εργασίας ε, είναι πολύ διαφορετικές και οι πολιτικές απασχόλησεις είναι πολύ διαφορετικές από χώρα σε χώρα. Και είναι πάντα αρμοδιότητα των κρατών μελών για το σημείο 22. Δεν είμαι σίγουρη ότι κάθε ε, περίοδος μαθητείας, κάθε στάζ θα πρέπει να είναι αμοιβόμενο. Και δεν μου αρέσει αυτή η λέξη κατάλληλο ή αξιοπρεπές. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ψύχηση για τα νομοθετήματα που θα υπάρξουν στον τομέα αυτό. Είναι πολύ γενικόλογες αυτές οι διατυπώσεις. Μιλάμε επίσης για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Και εδώ μπορεί να υπάρχουν ε, απλουστευτικές, απλουστευτικές ερμηνείες και γενικά σε πολλές νομικές ε, πράξεις, πολλά νομοθετήματα ε, λέμε ότι πρέπει να υποχρεωθούν τα κράτη να αναλάβουν δράση σε κάποιους τομείς κτλ. Αλλά καλύτερα να αναφερθούμε στην υπευθυνότητα των εργοδοτών και εργαζομένων. Αυτοί είναι οι παίκτες στην αγορά εργασίας. Αυτοί πρέπει να εφαρμόσουν ε, την οδηγία. Η ποιότητα της εφαρμογής είναι δική τους ευθύνη. Ίσως λοιπόν στα κείμενά μας να έπρεπε να τονίσουμε περισσότερο την ευθύνη εργοδοτών και εργαζομένων. Ο κύριος ε, Σίμον, Σάιμον αναφερόμενος στο σημείο 19 αναφέρθηκε στην αναθεώρηση της, ε, των κατεξοδότηση πράξεων που σχετίζονται με την οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων. Ο, ο πρόεδρος Γιούνκερ είπε ότι θα πρέπει να δούμε πώς εφαρμόζεται αυτή η οδηγία. Κατά την προηγούμενη θητεία εγκρίναμε την ε, εφαρμοστική οδηγία και θα πρέπει τώρα να δούμε πώς εφαρμόζεται. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πυρίνσκι. Ευχαριστώ. Στο σημείο 13 καλούμε την Επιτροπή επιγόντως να εξαιρέσει τις παραγωγικές επενδύσεις, για παράδειγμα για την εκπαίδευση, την έρευνα και την ανάπτυξη, από τους στόχους για το έλλειμμα που καθορίζονται με βάση τους νοσιακούς και εθνικούς νόμους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να διευκολύνουμε αυτό που πολλοί είπαν ήδη. Να υπάρξει απτή ανάπτυξη των επενδύσεων σε εθνικό επίπεδο. Για να ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη και την απασχόληση. Διότι το ευρωπαϊκό εξάμεινο, όπως λέγεται το σημείο 3, βασίζεται σε εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων και τους στόχους που θέτουν οι κυβερνήσεις και τους οποίους ε, εξετάζει και η Κομισιόν. Και υπάρχει περίπτωση λοιπόν να αποφασίσει η Κομισιόν ότι υπάρχει θέμα υπερβολικού ελλείμματος. Αν λοιπόν εγκρίνουμε αυτό το αίτημα, θα ήταν σημαντικό να υπάρχει αυτή η εξαίρεση, τώρα ακριβώς που τα κράτη-μέλη ε, εκπονούν τους προπολογισμού τους. Θα τους δώσει την αναγκαία ευελιξία για να αυξήσουν ε, τις επενδύσεις τους. Και αυτό ε, τίθεται στα πλαίσια του ευρύτερου θέματος της κοινωνικής συνοχής και της πολιτικής συνοχής που αναθεώρησε η Ένωση για την περίοδο 2014-2020. Σήμερα οι εκπρόσωποι της Κομισιόν στην Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής υπέβαλαν μια έκθεση που τονίζει ότι η πολιτική συνοχής είναι ένας από τους τρεις πυλώνες για να έχουμε ανάπτυξη, απασχόληση κτλ. Μαζί με την δημοσιονομική εξυγένση και τις διαφορετικέ μεταρρυθμίσεις. Η Επιτροπή λοιπόν επέμεινε ιδιαίτερα στο ότι η συνοχή θα πρέπει να φέρει επενδύσεις, χρηματοδότηση, ιδιαίτερα στις χώρες που έχουν μειώσει ιδιαίτερα τις δημόσιες επενδύσεις για να μειώσουν ε, το έλλειμμα. Η έκθεση λοιπόν αυτή και συμφωνώ με όσα υπόθηκαν για την ε, θαυμάσια ποιότητά της. Η έκθεση λοιπόν αυτή ξεκινάει λέγοντας στο α ότι οι ε, αποκλίσεις του επίπεδου των περιφερειών των κρατών μελών αυξάνονται. Οι ανισότητες και λέει επίσης περαιτέρω ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο μας έχει απομακρύνει από την επίτευξη των στόχων ε, των κοινωνικών και απασχόλησης ε, του θεματολογίου 2020. Εάν δεν αντιμετωπίσουμε τις διευρυνόμενες ανισότητες και τη στασιμότητα και τον αποπληθωρισμό ε, από τους οποίους ε, υποφέρει η ευρωπαϊκή οικονομία, όλα αυτά που θέλουμε είναι ανέφικτα. Γι' αυτό πιστεύω ότι η Επιτροπή μας θα πρέπει να έχει ως άμεση αποστολή να πείσει την ε, Οικονομική Επιτροπή ότι πρέπει να αλλάξει προσανατολισμό και να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτά που κάνουμε στο παρελθόν δεν έχει πλέον καμία έννοια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Τη Jane Collins. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τις προσπάθειες που κατέβαλε. Υπάρχουν όμως ένα-δυο σημεία που θα ήθελα να θέσω σε ό,τι αφορά το έγγραφο της Επιτροπής. Ενδεχομένως το πιο εντυπωσιακό σημείο είναι η παραγράφος 12 και το αίτημα να δαπανηθούν 300 δισεκατομμύρια ευρώ. Πραγματικά ένα αμύθιτο ποσό. Αυτό που θα ήθελα να γνωρίζω είναι από πού περιμένετε να προκύψουν αυτά τα 300 δις. Τα λεφτά δεν φυτρώνουν στα δέντρα. Θα πρέπει να προέρθει από τα χρήματα των φορολογούμενων, των φορολογούμενων που δίνουν αγώνα για να πληρώσουν αυτά που οφείλουν. Ενδεχομένω από τους ε, ε, συνταξιούχους θα κληθούν να πληρώσουν αυτό το λογαριασμό καθημερινοί άνθρωποι που δίνουν αγώνα για να επιβιώσουν. Κανένα στον πραγματικό κόσμο δεν ψήφισε Γι' αυτό και δαπανώνται, σπαταλώνται εκατομμύρια ε, κονδύλια. Η παράγραφος 19 ε, ζητά την πρόθεση της ελευθερίας κίνησης. Ε, αυτό τι σημαίνει, ανοίγουμε στις πόρτες τη μετανάστευση. Την τελευταία χρονιά η ιστοσελίδα ήταν η αιτία που πολλοί άνθρωποι χρειάστηκαν να μεταναστεύσουν. Εσείς λέτε ότι θα πρέπει να καταστήσουμε ευκολότερο για τους μετανάστες να έρθουν και να αναζητήσουν εργασία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Χρειαζόμαστε ελεγχόμενη μετανάστευση, να χρησιμοποιήσουμε το σύστημα των θεωρήσεων και των points της βαθμολογίας που χρησιμοποιούν στην Αυστραλία. Τέλος, θα ήθελα να τονίσω την παράγραφο, να αναφερθώ στην παράγραφο 19 που ζητάει ε, για ένα ελάχιστο ε, μισθό της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και για ε, νομοθεσία που θα εξασφαλίσει την ελευθερία διακίνησης. Ιδιαίτερα στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν άνθρωποι που είναι κατά αυτών. Ψήφισαν για λιγότερες δαπάνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για ε, πιο περιορισμένη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για, λιγότερες, ε, για λιγότερη εξουσία και για ένα λεγόμενο σύστημα μετανάστευσης. Ε, ευχαριστώ πολύ. Thank you, Mr. Ευχαριστώ, κύριος Λόπες. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Πολύ σύντομα να, συγχαρώ τον εισηγητή, τον Σέρχιο Γκουκέρ, για τη θαυμάσια εργασία του. Αυτό αποδεικνύει τις σημαντικές συζητήσεις θα έχουμε τα επόμενα χρόνια για τα οικονομικά θέματα, τις επιπτώσεις της οικονομίας, ιδιαίτερα στην αγορά εργασίας συμπτώσεις των πολιτικών της Ένωσης. Και τώρα που είδαμε τα πολύ άσχημα μακροοικονομικά δεδομένα για τον Αύγουστο και ολόκληρη την Ευρώπη, είναι πολύ επίκαιρο το θέμα αυτό. Αυτό αποδεικνύει όχι μόνο τις κοινωνικές επιπτώσεις, δηλαδή την κοινωνική ανισότητα, την έλλειψη κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά το ότι είναι και αναποτελεσματική από καθαρά οικονομική άποψη η πολιτική που ακολουθείτε σε σχέση με τα προβλήματα αυτές οι πολιτικές ε, λιτότητας, ε, εσωτερικής υποτίμησης, μείωση των μισθών για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και περιοριστική νομισματική πολιτική, αυτή ήταν η απάντηση που έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια στα προβλήματά μας. Αποδείχθηκε ότι είναι απόλυτα και αναπτολισματική και άδικη. Ιδιαίτερα όσον αφορά την αγορά εργασίας. Ιδιαίτερα. Μακροοικονομικά μειώνεται η εσωτερική κατανάλωση, κινητήριε δυνάμει όπως για παράδειγμα ε, ο δημόσιο τομέας για την οικονομία ε, χειραγωγούνται, μειώνεται η σημασία τους και δεν κερδίσαμε ανταγωνιστικότητα έναντι των ανταγωνιστών μας παγκόσμια, όπως αναγνώρισε και ο ΣΑ πρόσφατα. υπάρχουν τρομερές επιπτώσεις για τη φτώχεια. Όχι μόνο αυτή η εντύπωση ότι έχουμε πέσει σε, έχουμε πέσει μια άβυση από την οποία δεν μπορούμε να βγούμε, αλλά υπάρχει μια κατάσταση κοινωνικής ανισότητας που δεν την είχαμε ξαναδεί από το 19ο αιώνα. Αυτά είναι πολύ ανισχυτικά. Πρέπει λοιπόν να στείλουμε μια, ένα πολύ σαφές μήνυμα. Η οικονομική προσαρμογή δεν μπορεί να γίνει μόνο σε σχέση με την ε, προσφορά. Έχουμε κρίση και στη ζήτηση. Αν κάνουμε μόνο μέσω της μείωσης των μισθών προσαρμογές στην ζήτηση, τότε έχουμε πρόβλημα. Έχουμε κάποια μηνύματα από τον νέο πρόεδρο της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το σύνολο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του τελευταίους μήνες προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτές οι διακηρύξεις θα γίνουν πράξεις. Και όπως είπε μια, συντρόφ, μια σύντροφος, η δράση μας πρέπει να βασίζεται σε αξίες και σε ιδέες. Γιατί το ζήτημα δεν είναι να αποφασίζουμε γιατί χρώμα θα έχουν τα χαρτονομίσματα, αλλά να υπάρχει αξιοπρέπεια για όλους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Σκέλερ. I Απλώς θα ήθελα να μου πείτε το εξή. Αυτά τα τελευταία πενταετία επικρίσεις δηλαδή, πόσες τέτοιες ευέλικτες θέσεις εργασίας δημιουργήσαμε, γιατί πολλές φορές αυτές είναι αυτό το οποίο είναι ουσιαστικά η η θέση του εργαζόμενου ο οποίος πεινάει. Και έχουμε και αυτές τις ε, μητέρες που έχουν υποχρέωση τα παιδιά τους, πολλές φορές δηλαδή αυτές τις θέσεις προσφέρονται σε κάποιον που δεν τις χρειάζεται, δεν τις θέλει. Η Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε και τώρα να δώσουμε το λόγο στον κύριο Γιώτα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρόεδρε, έχετε το λόγο. Αξιότιμοι κύριε βουλευτέ, εμείς χαιρετίζουμε τη δεσμευσή σας για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Το Κοινοβούλιο έχει να διαρροντήσει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και εμείς παρακολουθούμε με προσοχή όλα αυτά τα οποία συστήνεται. Τη σημερινή μέρα, βέβαια, αυτό είναι ό,τι πιο σημαντικό και σήμερα. Ακριβώ από τη συζήτηση αναδεικνύεται το ότι θα πρέπει κάτι να γίνει, μια, το ότι έχουμε περίπλοκε ε, μπροστά μα ε, προκλήσει που έχει να με το η Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το 2014 αυτό το εξάμεινο ήταν το τέταρτο κατά σειράν και έδειξε ότι είχε αρχίσει να αποδίδει καρπούς, αλλά όχι επαρκώς. Και η αποτελεσματικότητα αυτού του εξαμένου εξαρτάται από την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων. Κάτι το οποίο είναι ένα σημαντικό στοιχείο, το οποίο θα καθορίσει τα αποτελέσματα. Πέρυσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεσήμανε ότι θα πρέπει να υπάρχει περισσότερη παρακολούθηση των μεταρρυθμίσεων, θα πρέπει να υπάρχουν συστάσεις σε κάθε χώρα χωριστά, θα πρέπει να υπάρχει επίσης με περισσότερη δημιουργούς χαρακτήρα υπάρχει με τα κρατημέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει από κοντά να παρακολουθεί την πρόοδο και την υλοποίηση σύμφωνα με τα όσα ορίζει η συνθήκη και το σύμφωνο σταθερότητα στο δε επόμενο εξάμεινο θα γίνει υπό την αιγίδα της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αν είναι Επιτροπή ε, έχει αναλάβει καθήκοντα τον Νοέμβριο. Προβλέπεται ο επόμενος κύκλος του επόμενου εξάμεινου να ξεκινήσει μετά κάποια στιγμή τέλο πάντων περί τα τέλη Νοεμβρίου όπως και τις προηγούμενες φορές. Οπότε και εμείς μελετήσαμε το σχέδιο κειμένου το δικό σας με μεγάλη προσοχή. Έχουμε κάποιες παρατηρήσεις και Περιμένουμε πώς και πώς να συνεργαστούμε στενότερα με τις πολιτικές ομάδες για να συζητήσουμε αυτές μας τις παρατηρήσεις. Ή Πρόεδρος, σας ευχαριστώ και τώρα να δώσουμε το λόγο για τις παρατηρήσεις του στον εισηγητή, τον κύριο Πριέτο, ούτως ώστε να ολοκληρώσει τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ όλους τους ε, συναδέλφους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα όσα είπανε όλοι αυτοί. Και τώρα έχει ξεκαταστεί για μένα τι πρεσβεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μίλησαν όχι μόνο όλες οι πολιτικές ομάδες, αλλά πάρα πολλοί συναδελφοί από όλες τις πολιτικές ομάδες. Νομίζω ότι υπάρχει μια γενικότερη συνένεση όσον αφορά την γνωμοδότησή μου, γιατί αυτό είναι κοινή επιθυμία. Πέραν της δικής μου άποψης, θέλουμε όλοι να υπάρξει ένα απτό σημαντικό αποτέλεσμα με μια τελική ψηφοφορία και έτσι να αντικατοπτρίζονται οι απόψεις μας γιατί πολλά θα διακυβευτούν και με την Οικονομική Επιτροπή αλλά και με τα θεσμικά όργανα της Ένωσης για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτούς τους σπουδαίους στόχους που είπαμε σε αυτή όλη την προβληματική. Αυτά που λέμε εδώ και τόσα χρόνια. Άρα να καταβληθεί προσπάθεια να έχουμε όλοι γενναιόδωρο πνεύμα για να φτάσουμε σε μια τέτοια ευρεία συνένεση που σχεδόν την έχουμε πετύχει. Με ειλικρίνεια, μόνο έτσι θα συνεχιστεί η συζήτηση έχοντας επίγνωση το ότι όταν μιλάμε για λιτότητα, όταν μιλούμε για λάθος συνταγές, πέραν δογμάτων, πέραν μηνυμάτων της πενταετίας που πέρασε, μιλάμε για για τον ε, σά, μιλάμε για φορείς ε, κοινωνικούς, μιλάμε για το δούνο του, ε, για ένα σώρο φορείς. Και έχουμε ακούσει ένα σωρό διαφορετικούς όρους, διαφορετικά ονόματα που βάφτισαν αυτή την λιτότητα. Οπότε υπάρχει αυτό το αυστηρότατο χρονοδιάγραμμα για την περικοπή των ελλημάτων, των στόχων Και τελικά τι γίναμε. Γίναμε οι πρωταθλητές της λιτότητας. Πέρασαν όλα αυτά τα χρόνια και με αυτές τις περικοπές φτάσαμε σε απίστευτες ανισότητες και φτώχεια. Και έτσι παρόλα αυτά μάλλον δεν έχουμε μπορέσει να ελέγξουμε ούτε το έλλειμμα ούτε το ποραπλασιαστικό αποτέλεσμα των δαπανών. Όχι. Δεν λέμε ότι δεν χρειάζεται καθόλου λιτότητα, αλλά όχι αυτή η υπερβολική, ακραία λιτότητα. Υποφέρει ο κόσμος. Δεν γίνεται τίποτα έτσι σε σχέση με το έλλειμμα. Και γι' αυτό και θέλουμε η Επιτροπή της Απασχόλησης να στείλει αυτό το μήνυμα τώρα που έχει φουντώσει η συζήτηση στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Και έτσι να μπορέσουμε να βρούμε τη σωστή δόση του φαρμακού. Να μην έχουμε αυτή την ακραία, αχαλήνωτη λιτότητα. Άλλωστε όλος ο κόσμος, όλα τα θεσμικά όργανα το επικρίνουν αυτό το φαινόμενο. Το είπε και η κυρία Κόλλιν. Πού θα βρεθούν τα χρήματα ούτω ώστε να γίνουν οι επενδύσεις. Μας έλεγε ότι θα βγουν από ένα κορδανά, θα βγουν από μια καταλήστευση των, ε, των πορτοφολιών του, του, του, του κόσμου. Όμως έχουμε αυτή την έκθεση ε, ας πούμε του Ινστιτούτου των Παρισίων και άλλων ανεξαρτήτων ε, ιδρυμάτων και λέει ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα καταπολέμησης του ελλείμματος πιο ευέλικτο και έτσι να μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε αυτά τα 85 ε, εκατομμύρια ετησίως από την Ευρωζώνη. Δεν χρειάζεται η αύξηση των φόρων, δεν χρειάζεται αυτού του είδους η, η ταλαιπωρία του κόσμου για να μπορέσουμε να πρικοδοτήσουμε τις ε, ε, επενδύσεις για να μπορέσουμε να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα της μείωσης του ελλείμματος. Άκουσα τι είπε και η κυρία Λόπεθ. Μας μίλησε για το για τον χρυσούν κανόνα, για την ε, κρατική πολιτική σχετικά με το έλλειμμα. Το θέμα είναι το πώς θα ευνοήσουμε τα θεσμικά όργανα, τους δημόσιους φορείς. Να υπάρχει ένας ενάρετος κύκλος που να οδηγήσει σε οικονομική ανάπτυξη αλλά και μεσοπρόθεσμα σε ισότητα ευκαιριών. Πάντα το λέγαμε. Υπάρχουν οι άλλες πολιτικές που βοηθούν. Πολιτική εκπαίδευση, ε, παραγωγικές επενδύσεις κλπ. Σε κάποιες χώρες μπόρεσαν οι ρυθμικά όργανα να κάνουν κάποιο είδους διάσωση. Αλλά πέραν του ελλείμματος να έχουν το, ένα καλύτερο ε, χρονοδιάγραμμα. Α πούμε έχουμε 40 δι στην Ισπανία όσον αφορά τη διάσωση. Δόθηκαν στις τράπεζες. Και είχαμε τέσσερι μονάδες λιγότερο έλλειμμα έτσι. Αυτό όμως δεν συνυπολογίστηκε. Τι έγινε με την παιδεία. Προχώρησαν στις περικοπές. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας λέει ότι είναι ανησυχητικό το ότι στα 25 κρατημέλη, έχουμε περικοπές στην παιδεία και έχουν παρόλα αυτά αυτές τις, τις περικοπές στην παιδεία. Αυτό δείχνει μια ασυνέπεια στην ιστορική μας λογική. Επομένως, αυτό θα πρέπει να τονίσουμε. Τελικά, για άλλη μια φορά, αυτό είναι θέμα πολιτικής βούλησης. επιτρέπεται αυτό με την σωστή χρήση και ερμηνεία των συνθήκων υπάρχει ευέλικτη ρύθμιση. Ήδη κάποιοι συνάδελφοι από εδώ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με κάποιου είδου αξιολόγηση όσον αφορά το, αυτό το, το πλάνο, το πρόγραμμα εγγύηση τη ε, απασχόληση των νέων. Αυτό γιατί ε, ανησυχούμε, δεν θεωρούμε ότι προχώρησε η υλοποίηση αυτού, αυτών των εγγύσεων για τους νέους τόσο γρήγορα και οδηγούμεθα σε κάποιες πολιτικές κρατών μελών που δεν είναι αποτελεσματικέ για να πολεμηθεί η ανεργία των νέων. Οπότε, τι γίνεται, απλώς υπάρχει κάποια μεταφορά πόρων. Δεν είναι αποτελεσματικό αυτό. Δεν θα πρέπει να προορίζονται αυτά τα χρήματα εκεί που δεν δημιουργείται κάποιο αποτέλεσμα. Αντίθετα, να χαράσσονται πολιτικές που να επιλύουν το πρόβλημα. Βεβαίω χρειάζεται ευελιξία. Και επομένω, ο Ευρωπαϊκό Κοροφανά να χρηματοδοτεί κάποιε πολιτικέ αποτελεσματικέ οι οποίε να δημιουργούν απασχόληση αξιοπρεπή. Και βέβαια να υπάρξει πολιτική βούληση αύξηση του κοινωτικού προπολογισμού. Και επίσης δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με πάρα πολλά από όσα είπαν οι προλαλήσαντες. Ότι δηλαδή θέλουμε να πετύχουμε τα μέσα που μένα χρόνια ποιοτικέ θέσει απασχόληση. Την επόμενη τετραετία αυτό θα πρέπει να γίνει και πώς θα συρρυκνώσουμε την ανεργία και την ανεργία των νέων. η ανεργία όλο ένα και περισσότερο γίνεται μια πραγματικότητα και οδηγεί σε αυτού του είδους την φτώχεια των εργαζομένων. Να μειώνεται η ανεργία, να βελτιώνεται η αγορά απασχόλησης, το οποίο εξαρτάται πάλι από πάρα πολλούς οι οποίοι δουλεύουν λίγες ώρες, δεν λαμβάνεται αυτό επαρκώς υπόψη και όπως είπε και η κυρία Μακεντάρη, οι επιχειρήσεις δημιουργούν απασχόληση. Όμως θα πρέπει να υπάρξει επαρκή νομοθετικό πλαίσιο, τόσο ώστε οι Ευρωπαίοι εργαζόμενοι να έχουν ισότητα ευκαιριών, γιατί όταν πριν από λίγους μήνες στην Ομοσπονδιακή Βουλή είπε η κυρία Μέρκελ ότι η ευελιξία δημιουργεί προβλήματα όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα. Έτσι, θα πρέπει οι εργαζόμενοι να σπαστούν το μοντέλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απασχόληση είναι πολύ περισσότερο από κάτι το οποίο απλώς κατοχυρώνεται από την νομοθεσία. Είναι κάτι το οποίο αποτελεί τον ομφάλιο λόρο της σύνδεσης του ατόμου με την κοινωνία. Άρα να διευκολύνουμε τις επιχειρήσεις για να δημιουργείται επασχόληση. Αλλά επίσης δεν θα πρέπει να αποκόπτονται οι εργαζόμενοι από την ε, κοινωνία αποστερώντας τους την αξιοπρέπεια που χρειάζεται προς τούτο. Επίσης, να μπει ένα τέρμα στις λαϊκιστικές φωνές με κάποιο είδους εθνικές ε, εκστρατείες που είναι άσχετες τελείως με αυτά που προτείνω εγώ στο κείμενο ή και είναι άσχετο με τα όσα πρεσβεύουμε οι περισσότερο στην Επιτροπή μας, κυρία Κόλλιντζ. Εγώ ως εισηγητής θέλω να δω πώς θα προσπαθήσουμε να έχουμε έναν ε, διάλογο που να σου οδηγήσει σε κάποιες ε, ισχυρές τοποθετήσεις και επιχειρήματα και να μην ε, όλοι σε κάποιο είδους ε, δημαγωγικές ε, ακρότητες. Εκμεταλλευόμενοι τον κόσμο που πάσχει τώρα από την κρίση. Εκεί διαφωνούμε. για αυτού του είδους. Δεν, μιλάμε τώρα για την μετανάστευση, για το θέλετε εσείς τώρα να συνδέσετε το Ιούρες με το θέμα της μετανάστευσης διαφόρων χωρών. Αυτό είναι ανησυχητικό, είναι δημαγωγικό, είναι κάτι το οποίο δεν έχει προηγούμενο στην εδώ, στην Επιτροπή μας. Έτσι συγχαίρεται τα πράγματα. Έτσι μπερδεύετε ή προσπαθείτε να μπερδέψετε τους συναδέλφους της Επιτροπής. Θέλουμε στην πράξη να έχουμε ενιαία αγορά εργασία στην Ένωση. Άρα θα πρέπει να προσφέρουμε κάποιες εγγύησει εργασία. Γιατί η κοινή αγορά και η νέα αγορά δεν πάνε να πει μόνο ελεύθερη διακίνηση. Χρειάζονται και εγγύησει που να βοηθούν την κινητικότητα. Σε αυτό αποσκοπεί το έωρε. Θα πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί. Εντάξει, δεν λέω να, να μεταρρυθμιστεί αν χρειάζεται. Οπότε, η εγγύηση κάποιων προϋποθέσεων, αξιολόγηση, να δούμε τι προβλήματα χρειάζονται και να μεταρρυθμίσουμε. Αλλά δεν μιλάμε τώρα μόνο για τους ε, μετανάστες των τρίτων χωρών μιλούμε, για τους Ισπανούς που θα πάνε στη Γερμανία, για τους Πορτογάλους που θα πάνε αλλού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε αυτούς θα πρέπει να παράσχουμε εγγύησεις ενίας αγοράς που πάει να πει ευρωπαϊκή οικοδόμηση. Τέτοια Ευρώπη θέλουμε. Πέραν των ευκόλων κραυγών και επιχειρημάτων στην πράξη θέλουμε να το κάνουμε αυτό. Δεν θέλω λοιπόν να ολιστήσουμε σε κάτι τέτοια επιχειρήματα στην Επιτροπή μα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους σας για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Προθεσμία, κατάθεση τροπολογιών 9 Σεπτεμβρίου. Η επόμενη συνάντησή μας, οι τροπολογίες μπορούν να κατατεθούν μόνο στα αγγλικά. Γιατί υπάρχει πρόβλημα χρόνου. Η επόμενη συνάντηση της Επιτροπής προβλέπεται για τις 29 Σεπτεμβρίου θα τα πούμε τότε. Σας ευχαριστώ πολύ.